Ωραία, να ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Να σας ενημερώσω συγκεκριμένα για τις αποφάσεις των συντονιστών. Λοιπόν, θα κάνουμε μία γνωμοδότηση. Η κυρία Πρόεδρος συγκεκριμένα θα κάνει μία γνωμοδότηση για την ε, επιτήρηση της εφαρμογής της ενωσιακή νομοθεσίας. Συζητήθηκαν επίσης πέντε συγκεκριμένες αναφορές σήμερα το πρωί. Η 624 θα παραμείνει ανοιχτή. Η 690 θα γίνει δεκτή. Και, και για την 676, την 680 και την 682 οι συντονιστές αποδέχτηκαν τις προτάσεις της Προέδρου. Όσον αφορά την έκθεση για το πρόγραμμα εργασιών της ΤΟΑ για το 2018 εγκρίθηκε και επ' αυτού η πρόταση της Προέδρου. Και όσον αφορά το χτένισμα των παλιών αναφορών αναβλήθηκε η εξέτασή του για τον Ιανουάριο. Η έκθεση της 22 Νοεμβρίου θα αναβληθεί επίσης για τον Ιανουάριο. Και, και η αναφορά 1012 θα μας απασχολήσει το Φεβρουάριο. Θεωρείται αποδεκτή και θα μας απασχολήσει το Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ε, μόλυνση των υδάτων στην Λουσατία. Αυτά μου ζήτησε η κυρία Πρόεδρος να σας ε, πω. Και τώρα να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Περνάμε τώρα στην πρώτη αναφορά που θα μας αποσχολήσει σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για ένα Ρουμάνο πολίτη, ο αναφέρον ε, Ρουμάνος, για τον ε, μη σεβασμό μίας οδηγίας και θα δώσω το λόγο ε, στον αναφέροντα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής ε, Αναφορών. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ε, μιλήσω. There is a Okay, but there is no translation to other languages. I wait. Is it okay? Now? No, Υπάρχει μετάφραση τώρα. Again, excuse me, please. Okay, no problem. So. Ωραία, ευχαριστώ. Ε, αξιότιμη Επιτροπή Αναφορών, σας ευχαριστώ για την ε, αποφασιστικότητα με την οποία με αντικειμενικό τρόπο σας παρουσίασα την αρχική μου αναφορά. Οι ρουμανικές αρχές αναγνώσαν τις σοβαρές αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας 2014-42 κάθετος ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το μη σεβασμό των ε, προθεσμιών για τη μεταφορά από τις 4 Οκτωβρίου 2016. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι μέχρι τώρα, 28 Νοεμβρίου 2017, δεν έχει γίνει τίποτα για τη μεταφορά των δικονομικών εγγυήσεων όσον αφορά μια δίκαιη δίκη όπως καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και από τις παγκόσμιες προδιαγραφές, το άρθρο 8 της οδηγίας στην οποία προαναφέρθηκα. Ενώ η τιμωρητική πλευρά της οδηγίας μεταφέρθηκε στην ρουμανική νομοθεσία εγκαίρως για τις δικονομικές εγγυήσεις ε, και για την ισότητα δυνατοτήτων η Ρουμανία έκανε μόνο διακήρυξεις και εξακολουθεί να κάνει το ίδιο. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή είναι ένα καταρρεύσαν ευρωπαϊκό κράτος όσον αφορά τις ε, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προδιαγραφές για τις, ασφα... για τις ε, δημόσιες ελευθερίες. Η Ρουμανία είναι καταπιστικό κράτος και καταπιέζει τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της. Το γεγονός ότι δεν μετέφερε αυτή την οδηγία στο σύνολό της εσκεμένα αγνοώντας τις δικονομικές εγγυήσεις για να μπορέσει να γίνεται ε, αποτελεσματική υπεράσπιση είναι απομάκρυνση από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε όταν ενετάχθηκε στην Ένωση. Έτσι λοιπόν οι καλές προθέσεις αυτής της οδηγίας θεωρούνται από τους πολίτες της Ρουμανίας ως υπερβολικά τιμωρητικές και καταχρηστικές, ενώ στην ουσία η οδηγία είναι ισορροπημένη και δίκαιη η στρέβλωση των στόχων της ε, οδηγίας στην ουσία καταδεικνύει και τα θετικά της και στρέφεται μια τέτοια εφαρμογή κατά των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ουσία έτσι ενισχύεται ο ευρωσκεπτικισμός. Γι' αυτό τον λόγο η αντίδρασή σας πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική. Να καταδείξετε την πραγματικότητα. Η απόφασή σας θα σας κάνει να προσεγγίσετε τους καταπιεζόμενους Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα η ρουμανική εφορία αφαιρεί τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών μόνο με υποθέσεις ότι είναι προϊόν εγκλημάτων και δεν έχουν καμία δυνατότητα να προσφύγουν οι πολίτες. Για παράδειγμα με την απόφαση 1207 κάθετος α κάθετος 2014 που ε, ανακοινώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014 από το ε, εφετείο του Βουκουρεστίου στην απόφαση 3694 κάθρος 3 2005. Στη Ρουμανία του 2017 η υψηλότερη μορφή της εθνικής δικαιοσύνης το ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο δεν αναγνωρίζει τα μέτρα της οδηγίας αυτής άρα δεν υπάρχουν προδιαγραφές δίκαιης δίκης ενώ θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί πριν από 12 μήνες. Παραθέτω την ε, ποινική απόφαση 199 κάθος 2017 που ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 από το Ανώτατο Αναρετικό Δικαστήριο στην υπόθεση 4031 κάθος 1 κάθος 2016. Επειδή η έφεση βασιζόταν σε κανόνες που δεν αναγνωρίζει η ποινική δικονομία, το ανώτοτο δικαστήριο την απορρίπτει. Φασίστηκε στο άρθρο 8, παραγράφους 6 και 7 της Οδηγίας 2014-42 κάθος Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρθηκαν αποδεικνύουν ότι υπάρχει κατάχρηση, όπως έλεγα και στην αρχική μου αναφορά. Το γεγονό ότι δεν υπάρχουν δικονομικές δικαιοσύνης μετατρέπει οποιαδήποτε αστική ή ποινική απόφαση σε καταχρηστική μπορώ να σας ε, γνωστοποιήσω τις αποφάσεις αυτές όποτε θέλετε. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλετε και θεωρώ ότι οι άσκοπες και λαθασμένες αντιδράσεις των ρουμανικών αρχών πρέπει ε, να αντιμετωπιστούν για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών που πρέπει να βασίζονται στο τεκμήριο αθωότητας και σε ουσιαστικές δυνατότητες έφεσης. Προς το παρόν πρέπει να συνεχίσουμε τις διαδικασίες επί παραβάσεις να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Επί συγγνώμη. Από αυτήν την πλευρά η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να θεωρήσει ότι η καθυστέρηση στην μεταφορά στη ρουμανική νομοθεσία αυτής της οδηγίας έχει ουσιώδη αποτελέσματα. Στο σύνολό τη βεβαίω στην μεταφορά τη οδηγία. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει στα περαιτέρω βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επί παραβάσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρου Μαριάννη Ιάνκου, εκπροσωπούμενος από τον Αλεξάνδρου Εμιλιάν Ιάνκου. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Σεμπαστιάν εκ μέρους της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα που επισημαίνει αυτή την υπόθεση στην Επιτροπή μας. Αναφερόμαστε στην οδηγία περί κατάσχεσης ε, ε, περιουσιακών στοιχείων από προϊόντων εγκλήματο. Ε, που είχε η ημερομηνία μεταφορά το 2016, όπως πολλά κράτη-μέλη, η Ρουμανία πριν από την προθεσμία μεταφοράς έστειλε τις σημερινές τους διατάξεις, αυτό που έχουν ήδη στον ποινικό τους κώδικα, ε, στην ποινική του οικονομία περί κατάσχεσης τον Ιούνιο του 2000, τον Ιούλιο του 2016 και μας ανέφεραν ότι αυτή η ειδοποίηση δεν θα είχε ολοκληρωθεί αλλά ότι περαιτέρω νομικές διατάξεις ήταν απαραίτητες για πλήρη ευθυγράμμιση της ρουμανικής νομοθεσίας με την οδηγία. λόγω έλλειψης περαιτέρω μέτρων ε, ε, το 2016 δεν κοινοποιηθήκαν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ανέλαβε δράση με επίσημη ε, επιστολή προς την ρουμανική κυβέρνηση για μη κοινοποίηση των υπόλοιπων διατάξεων. Η διαδικασία παραβάση έχει ανοίξει από το Νοέμβριο του 2016. Μετά από αυτό έχουμε μείνει σε επαφή με τη ρουμανική κυβέρνηση για να μάθουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά τους για πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Έχουμε λάβει τις πληροφορίες ότι τον Αύγουστο η ρουμανική κυβέρνηση έστειλε το νομοσχέδιο στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και δημόσια διαβούλευση. Και δεν έχουμε μάθει τίποτα νεότερο. Από ό,τι γνωρίζουμε, ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα ενώπιον τη ρωμανική κυβέρνηση. Από όσο γνωρίζουμε από πλευρά Κομισιόν, φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση και αναμένουμε ε, κοινοποίηση από την ρωμανική κυβέρνηση μόλις το νομικό αυτοκείμενο υιοθετηθεί, ώστε να ελέγξουμε κατά πόσο το κείμενο του νομοθετήματος μεταφέρει πλήρως τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ωραία λοιπόν, τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας τα όσα είπε η Κομισιόν, πρέπει να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η νομοθεσία αυτή οθετήθηκε τον Αύγουστο του 2017. Ενώ ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας λέει ότι δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί. Λοιπόν, η νομοθεσία έχει εγκριθεί, έχει υιοθετηθεί λίγο αργότερα τον Αύγουστο του 2017 και η θέση της ομάδας μας είναι να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να δει κατά πόσο η μεταφορά έγινε σωστά. Ωστόσο, για να μπορούμε εμεί να πραγματοποιήσουμε αυτή την, αυτόν τον έλεγχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει στα χέρια τη ε, έγκυρε πληροφορίε. Αν όμω η Κομισιόν έρχεται και μα λέει ότι δεν έχει λάβει τέτοιε πληροφορίε, εκεί έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη αυτές τις πληροφορίες και ελέγξτε κατά πόσο έχει γίνει σωστά η μεταφορά στη ρουμανική νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά μέχρι ότου βεβαιωθούμε ότι υπήρξε μεταφορά. Όσον αφορά τις, άλλες, ε, τις δύο άλλες αναφορές, ε, ο κύριος Γιάρ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το λόγο γιατί εγώ θα πρέπει να πάω να, φυ... να αναχωρήσω από την αίθουσα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέντα. Να ρωτήσω τον κύριο Τίνες, θέλετε να απαντήσετε ή να αντιδράσετε στα όσα υπόθηκαν μόλις, όχι. Ναι, βάσει των όσων υπόθηκαν ε, έλαβε ο Αντιπρόεδρος ε, κ. Τίμερμανς ε, από τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μια επιστολή. Αυτό που υιοθετήθηκε ήταν η απόφαση της ρουμανικής κυβέρνησης να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο και να σταλεί στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο προσυζήτηση και έγκριση. Αυτές τις προφορέ λάβαμε εμείς. Δεν έχουμε λάβει κάτι, οτιδήποτε άλλο μετά από αυτό, από τη Ρουμανική κυβέρνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί το νομοσχέδιο ενώπιον του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Ε, αν υπήρξαν περαιτέρω εξελίξει ε, σε μεταγενέστερο στάδιο, η Κομισιόν δεν έχει ενημερωθεί. Ε, ευχαριστούμε. Αναφέρον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Όπως λέω και στην ομιλία μου, η οδηγία υλοποιήθηκε μόνο μερικώ. Κατά τη ραψή μου μόνο η κατασταλτική πλευρά, η τιμωρητική πλευρά. Έγινε κατάσχεση, για παράδειγμα, ήδη στην επιχείρησή μου, χωρίς να μου δοθεί ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας. Ναι, η οδηγία μένα έχει μεταφερθεί στην νομοθεσία, αλλά μόνο εν μέρη. Μόνο ε, το τιμωρητικό κομμάτι και πιστεύω ότι μια δημοκρατική χώρα, η ε, Ρουμανία που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μεταφέρει και να υλοποιεί πλήρω την οδηγία παρέχοντας και στις δύο πλευρές την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ε, στη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μου δεν εκλείσαν ποτέ στα δικαστήρια να υπερασπιστούν τι υποθέσει αυτέ. αλλά στο μεταξύ του τελευταίου μήνε έγινε ήδη κατάσχεση των δικών περιουσιακών στοιχείων βάσει υποθέσεων Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας προτείνω την εξής λύση. Είναι απόλυτα προφανές ότι η Ρουμανία φέρει ευθύνες, ε, έχει δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό η Ρουμανία έχει μεταφέρει την οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε το εξή. Ή θα αφήσουμε, ανοιχτή, θα αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά αναμένοντας νέες πληροφορίες. Αν συμφωνείτε, ας ε, προχωρήσουμε έτσι. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη αναφορά. Αναφέρον είναι ένας, ε, ένα άτομο ισπανικής ηθαγένειας σχετικά με το κόστος και την υποχρέωση παράσταση δικηγόρων σε ακροματικές διαδικασίες. Δεν είναι παρόν, οπότε θα δώσω το λόγο σε αυτόν που θα συνοψίσει την αναφορά. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο αναφέρον αναφέρεται στο επάγγελμα του προκουραδόρ, είναι κάτι ιδιαίτερο στην Ισπανία, όχι στο επάγγελμα του δικηγόρου, που στα ισπανικά ονομάζεται αμπογάδο. Ο αναφέρον εξηγεί ότι η υποχρέωση να, να χρησιμοποιείται προκουραδόρ στο δικαστήριο και οι ε, προαποφασισμένες τιμές ε, για αυτό ε, παραβαίνει την οδηγία 123 του 2006. Το επάγγελμα του προκουραδόρου υφίσταται μόνο στην Ισπανία και καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση με την τεχνική αντιπροσώπευση ε, των διαδίκων στο δικαστήριο δραστηριότητε ε, που σε άλλα κράτη-μέλη ε, είναι αρμοδιότητα δικηγόρου, καθώς επίσης και ε, καθήκοντα εφαρμογής και ενημέρωση επίδοσης εγγράφων που σε άλλα κράτη εκτελούνται από δικαστικούς επιμελητές ή από το δικαστήριο το ίδιο. Οι προκουραδόρες ε, υπογράφουν ε, έγγραφα εκ μέρους του πελάτη τους, τα υποβάλλουν στο δικαστήριο, ενώ οι δικηγόροι δίνουν νομικές συμβουλές και συνδρομή στους διαδίκους. Σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία γύρει ο, αναφέρον, ε, η Κομισιόν θα ήθελα να εξηγήσει το εξής. Έχουμε λάβει ε, ε, παράπονα για αυτό το θέμα και έχουμε έρθει σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές. Μάλιστα ξεκινήσαμε διαδικασία παραβάση για διάφορα θέματα με εξεταξή αυτών αυτά τα οποία αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά. Η Κομισιόν έστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2016. Οι Ισπανικές Αρχές επάντησαν το Φεβρουάριο του 2017 και αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες Κομισιόν αξιολογούν αυτή την απάντηση παρόλο ότι η διαδικασία παραβάση εκρέμει, θεωρούμε ότι είναι σωστό να περιμένουμε το αποτέλεσμά της πριν απαντήσουμε στην αναφορά. Ευχαριστώ. Peter Ο κύριος Γιάρ. Sí, yo creo... Όχι, η κυρία Σταράς. Ε, η Κομισιόν έδωσε τη σωστή απάντηση. Είπε ότι ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση. Αυτή τη στιγμή ανταλλάσσουν πληροφορίε με την Ισπανική κυβέρνηση και λέει ότι πρέπει να περιμένουμε. Οπότε α κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά για να δούμε ποια θα είναι η εκβασή τη ε, διαδικασία επί παραβάση και τη ανταλλαγή πληροφοριών. Ο κ. Γιάρ. Πολύ σωστή σύνοψη και συμφωνώ με την κυρία Σταράς. Ωραία, πρόεδρος. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε το θέμα. Ε, συμφωνούμε με την Κομισιόν, θα περιμένουμε την απάντηση της Ισπανικής κυβέρνησης και θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι τότε. Ωραία. Περνάμε στην επόμενη αναφορά. Πρόκειται για δύο συναφείς αναφορές, η, την 1523 του 2014 και την 512 του 2012. Πρόκειται για δύο Γερμανούς πικόους. Οι δύο αναφέροντες δεν είναι παρόντες από όσο γνωρίζω, οπότε θα ζητήσω από την, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να μας συνοψίσει ε, την άποψή της Κομισιόν. Yes, uh, Αυτές οι δύο αναφορές ε, αφορούν τη διαδικασία μικρών διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αδυναμίες στην ε, εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Εκεί τελειώνουν οι, ε, τα κοινά σημεία αυτών των δύο αναφορών, οπότε θα τις δούμε μία-μία. Πρώτη αναφορά, η 1523 του 2014 του κυρίου έχει μια δικαστική απόφαση και θέλει να την εφαρμόσει στην Ισπανία. Η εφαρμογή της απόφασης ε, δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαθέτουμε, του ζητήθηκε από το Ισπανικό Δικαστήριο, το οποίο είχε δεκτεί προηγουμένως την εφαρμογή, το εκτελεστό της απόφασης στην Ισπανία, του ζήτησε να αναφέρει αναφέρει το προσωπικό στοιχείο επί του οποίου θέλει να εφαρμοστεί η απόφαση. Αυτό είναι η τελευταία πληροφορία την οποία είχαμε λάβει, δεν ξέρουμε τι συνέβη αργότερα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία μικρών διαφορών, όπως και οποιαδήποτε άλλη δικαστική διαδικασία, εγγυάται μία απόφαση, αλλά όχι την, ε, την εκτελεστότητά της, την εκτέλεσή της. Και ε, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο κανονισμός καλύπτει όλες τις αστικές διαφορές και διασυνοριακά. Δηλαδή την, την ε, αναγνώριση μιας απόφασης ενός δικαστηρίου, ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος. Όμως σύμφωνα με τον κανονισμό η εκτέλεση της ίδιας της απόφασης ε, αποτελεί αντικείμενο της εθνικής νομοθεσίας του κράτους όπου γίνεται η εκτέλεση. Πάβει να είναι δηλαδή ευρωπαϊκό ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ισπανικές αρχές αναγνώρισαν πως πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση και ξεκίνησαν εθνικές διαδικασίες ε, εκτέλεσης. Λυπάμαι που αυτό απέτυχε, αλλά δεν έχουμε νομική βάση πάνω στην οποία να στηριχτούμε για να... Ε, παρέμβουμε ενώπιον των Ισπανικών αρχών. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία θεωρεί ότι αυτή η απόφαση είναι σαν να ήταν απόφαση που έχει εκδοθεί από Ισπανικό δικαστήριο και απαιτεί ακριβώς τα ίδια πράγματα που θα απαιτούσε αν η απόφαση ήταν από Ισπανικό δικαστήριο. Μπορεί πράγματι να είναι πιο δυσχερής η εκτέλεση στην Ισπανία, αλλά αυτό δεν αποτελεί ε, κομμάτι της διαδικασίας των μικρών διαφορών ε, και του κανονισμού. Οπότε, επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε παράβαση του κανονισμού Ευρωπαϊ... Ε, Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικρών Διαφορών εκ μέρους των Ισπανικών Αρχών. Η επόμενη περίπτωση είναι διαφορετική. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα δικαστική απόφαση, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε κάποια δικαστική απόφαση. Ο ένας Γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος εμπορεύεται τα προϊόντα του σε όλη την Ευρώπη παραπονιέται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με την εφαρμογή της διαδικασίας μικρών διαφορών. Δυστυχώς δεν υπέβαλε κανένας είδους έγγραφο που να τεκμηριώνει τους του. Οι ισχυρισμούς του, οι ισχυρισμοί του είναι λίγο δυσνόητη. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υφίστανται σε κάποια κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη γενικότερα σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας. Και χρειάζεται μια διδακτική δράση, ε, χρειάζεται να συνηθίσουν στη διαδικασία κλπ. Αλλά ποτέ δεν έχουμε δει ε, κάποιο δικαστήριο να αφιβάλλει για την ταυτότητα του ενάγοντος. για του αναγόμενου εντάξει, αλλά του ανάγοντα ποτέ. Ε, είναι θέμα βέβαια δικονομ, εθνικής δικονομίας αυτό. Ε, δυστυχώς εξαιτία της του περιορισμένου ε, χρονικού ορίζοντα ε, ο αναφέρον μας απάντησε ότι δεν έχει ε, τεκμηρίωση. Αναφέρει κάποια διαδικαστικά θέματα σε άλλα κράτη-μέλη, τη Γαλλία, τη Φιλανδία κλπ. Και πάλι χωρίς να μας υποβάλει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, απόδειξη ή κάποια δήλωση, επίσημη δήλωση. Έχουμε την εντύπωση ότι η πρόθεση του αναφέροντος είναι να μας επιστήσει την προσοχή στα πρακτικά προβλήματα προκειμένου να πάρουμε να αναλάβουμε δράση, το οποίο σε οριζόντιο επίπεδο το κάνουμε και είμαστε πάντα πρόθυμοι να το κάνουμε. Όμως δεν έχει κάποια διεκδίκηση. Επιπλέον αναφέρεται στο γερμανικό ε, στη γερμανική εντολή πληρωμής, διαδικασία εντολής πληρωμής ε, ως τρόπο ανάκτησης ποσών. Ε, η διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος πληρωμής που εφαρμόζεται τα τελευταία δέκα χρόνια βασίστηκε ακριβώς στο γερμανικό αντίστοιχο μοντέλο. Όλες αυτές οι πληροφορίες ε, βρίσκονται στο πόρταλ της Κομισιόν για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Εκεί περιλαμβάνονται όλες οι, ε, όλα τα ε, έγγραφα τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν, να σταλούν, να μεταφραστούν και ε, αναφέρονται και οδηγίες για την εφαρμογή της ε, διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό μικρών διαφορών, αυτός ε, πρόσφατα αναθεωρήθηκε και η αναθεώρησή του ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή. Και από ό,τι φαίνεται η διαδικασίες πηγαίνουν καλά, εφαρμόζονται γενικά οι αποφάσεις, δεν υπάρχουν οριζόντες και γενικευμένες αδυναμίες. Αυτά έχω να πω μόνο. Ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας να αναφερθώ σε μία μελέτη της Κομισιόν ότι η Κομισιόν εντόπισε τις κύριες αντιστάσεις. Πρώτα απ' όλα ε, οφείλονται σε άγνοια της ίδιας της διαδικασίας και το απρόβλεπτο κόστος και ο χρόνος που χρειάζεται για να επιδιωχθεί η πληρωμή μικροδιαφορών, η ρύθμιση. Θα αναφερθώ στην περίπτωση Βέλμπροκ. Οι αποφάσεις τις οποίες αναφέρεται είναι από το 2012, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια ο κύριος Βέλμπροκ. Ήδη το 2012 απευθύνθηκε εγγράφος προς τα, ευρωπαϊκά, προς τα ισπανικά δικαστήρια και κατόπιν ε, περνάει ένα γολγοθά ε, δεν τον ε, κολλησιεργούν του ζητάνε λοιπόν 50 ευρώ για το κόστος της ε, έφεσης ε, μετά φαίνεται ότι δεν ε, σημειώθηκε σωστά ότι λήφθησαν τα χρήματα του ξαναζητάνε εγώ θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ταχύτερη και φθηνότερη για την ρύθμιση μικροδιαφορών Καταλαβαίνω αυτά που είπατε, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας λέτε δηλαδή ότι εντάξει εφόσον είναι μέσα στην ισπανική μηχανή το θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή οποιοδήποτε ζητάει στην Ισπανία να εκτελεστεί μια απόφαση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται όπως ο αναφέρον. Και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να μάθουμε εάν έχουν υπάρξει επιτυχείς εκτελέσεις αποφάσεων στην Ισπανία. Από Ισπανούς ή από αλλοδαπούς. Και αν υπάρξει διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε ε, να κάνουμε να το βελτιώσουμε. Και το δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά ε, ε, οφείλονται μόνο σε γλωσσικές δυσχέρειες. Εγώ ντρέπομαι ενώπιον αυτού του αναφέροντος. Γράφει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καναλτών στο Κίελο και αυτοί γράφουν στον ε, χρεώστη και πληρώνει τουλάχιστον το κεφάλαιο. Δεν το έκανε ούτε ο κύριος Βίλαντ, ούτε η κυρία Βίξτρομ, η οποία έλαβε διάφορες επιστολές. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Δεν το έκανε το Ισπανικό Δικαστήριο. Το έκανε ένας φορέας ε, καταναλωτών, ο οποίος απλώς απευθύνθηκε στον, ε, στον χρεώστη. Αν ε, καταλάβουμε ότι ενώ στην αρχή οι πολίτες ε, ήταν πολύ ικανοποιημένοι που υπάρχει αυτή η διαδικασία επίλυσης μακροδιαφορών, αλλά όταν μετά διαπιστώσουμε ότι όταν πάει να εφαρμοστεί υπάρχουν τότιες, ε, τέτοιες διαδικασίες, τότε ως νομικός μπορώ να σας πω ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να υποσχόμαστε στους πολίτες πράγματα τα οποία δεν μπορούμε μετά να εφαρμόσουμε. Πρέπει να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να υπάρχει διάκριση εναντίον κανενός, αλλά θα πρέπει, εφόσον τα κράτη-μέλη έχουν τα ίδια συμβάλει στην έγκριση αυτών των διαδικασιών, να μην κοροϊδεύουν μετά τον κόσμο. Και να ξοδεύει ο κόσμος τόσα λεφτά και να κινείται σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει κανένα δίκαιο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αιτιολογημένο να πούμε ότι εφόσον είναι δίκαια αυτά τα αιτήματα δεν είναι τρόπος να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει ίσως να το μελετήσουμε περαιτέρω και να πούμε ότι η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Η καθυστέρηση του δικαίου είναι άρνηση δικαίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βίλαντ. Οπότε, να θέσω το εξή ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε καμία πρόταση. Κάνετε μία ανάλυση με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Λάξω προσεκτικά και τον κύριο Γκέρσκα και είπε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ότι η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Καλά σας κατάλαβα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα για να κάνει κάτι από αυτού. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι αρμοδιότητα των Ισπανικών αρχών. Οπότε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Δηλαδή το να επιδιώκουμε δίκιο και να επέρχεται αδικία είναι διαφορετικά πράγματα, όπως λέει και ο λαός μας. Μπορούμε και να το βάλουμε στο αρχείο το θέμα να πούμε ατυχία. Η διαδικασία στην Ισπανία έτσι είναι. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, που θα πρέπει να κάνουμε, είναι να στείλουμε μια επιστολή που να εκφράζει σαφώς ε, την ε, δυσαρέσκειά μας έναντι των ε, δραστηριοτήτων των Ισπανικών αρχών. Αυτός ο νόμος θέλει να προστατεύσει τα μικρά άτομα. Κοιτάξτε, Εάν υπάρχουν πολυεθνικές που θέλουν εκατομμύρια να εισπράξουν, τότε θα τα εισπράξουν. Υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που θα κάνουν ό,τι πρέπει για να τα εισπράξουν. Αλλά αν είναι ένα κάποιος ένας ε, μικρο... ένας πολίτης, ο οποίος έχει ένα μικρό συμφέρον και θέλει να τα εισπράξει, εσείς ή εγώ, και είναι νομικά όλα άρεστα, Αλλά δεν παίρνει τα χρήματά του. Μπορούμε να πούμε καλά ατυχία. Όπως είπε και ο κύριος Βίλαντ, ε, εν μέρη πήρε κάποια λεφτά λόγω της ε, επέμβασης αυτού του κέντρου καταναλωτών. Κοιτάξτε, θα έπρεπε να πούμε σαφώς στις ισπανικές αρχές ότι δεν είναι πράγματα αυτά. Να τους ρωτήσουμε, είστε εσείς ικανοποιημένοι με αυτή τη διαδικασία, σας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο πολίτης ε, πάει μπρος και πίσω και δεν επιτυχάνει τίποτα και περιμένουμε τελικά να κουραστεί και να εγκαταλείψει. Κάποια στιγμή θα εγκαταλείψει. Δεν είναι πράγματα αυτά. Χάνουμε κάθε αξιοπιστία. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε στον αναφέροντα όλα σωστά γίνανε, απλώς τα χρηματάζουν, δεν θα τα πάρεις. Είναι αυτό που λένε η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε να τους γράψουμε μια σαφή επιστολή που να τους πούμε ότι θέλουμε μια σαφή εξήγηση. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Και ίσως κάτι να προκύψει. Κάτι, κάτι να προκύψει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, συγκεκριμένη πρόταση, την οποία υποστηρίζω. Δηλαδή, θα αποστείλουμε μια επιστολή στο Ισπανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιστήσουμε την προσοχή τους επί των προβλημάτων που υπάρχουν στη διαδικασία από ό,τι φαίνεται και θα τους ζητήσουμε να ασχοληθούν με αυτό το θέμα σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία. Η πρότασή μας λοιπόν είναι επίσης να στείλουμε και μία επιστολή στην κυρία Γιούροβα για να επιστήσουμε την προσοχή της στο άλλο θέμα ότι δεν υπάρχουν ε, υποχρεωτικές υποχρεωτικές ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μία απόφαση που λαμβάνεται σε ένα, ευρωπαϊκό, σε ένα κράτος μέλος δεν ισχύει στα άλλα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτό το νομοθετικό κενό. Αυτή είναι η πρότασή μου. Λοιπόν, η 1053 κάθος 14, η αναφορά Βελμπρόκ θα παραμείνει ανοιχτή, ενώ οι άλλοι θα κλείσει. Εντάξει, ωραία. Επόμενη αναφορά. Είναι μια αναφορά που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Βίλαν. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θελήσαμε στις διαδικτυακές ε, πωλήσει και αυτός ο εικονικός κόσμος ε, ε, να διαπιστώσουμε και αυτός ο εικονικό κόσμος είναι διαφορετικός στον πραγματικό. Εάν κάνω μια αγορά στο ίντερνετ, έχω περισσότερα δικαιώματα από ε, έναν αγοραστή που πηγαίνει σε ένα μαγαζί. Αν πάω σε μια διαδικτυακή επιχείρηση, αγοράζω ένα ποτήρι που λέει ότι μπορεί να μπει στο πλυντήριο πιάτων και κύριε της Επιτροπής. Κύριε της Επιτροπής, σε, ε, σας αφορά αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, ε, τότε μπορώ να προσφύγω. Εάν το έχω αγοράσει επιτόπου στο, σε ένα ελληνικό νησί αυτό το ποτήρι, πρέπει να πάω σε αυτό το ελληνικό νησί για να απαιτήσω να επιστραφεί. Ενώ, εάν το έχω αγοράσει στο ίντερνετ, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Δεν ε, έχω διαβάσει την αναφορά. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να την κλείσουμε. Αλλά θα ήθελα οι κύριοι της Επιτροπής να λάβω μία απάντηση. Νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο. Και η πρότασή μου θα ήταν να προσπαθεί όταν υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, μεταξύ διαφόρων κρατών να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, θέσεις που να ασχολούνται με αυτά τα θέματα και να επιβάλλουν την εκτέλεση. Θα έπρεπε η Κομισιόν να καταλάβει τη φύση του προβλήματος που είναι φανερό ότι υφίσταται. ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ιδέα είναι άριστη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο θα θέλαμε να αναλάβουμε αυτή τη δράση θα μας ρωτήσει με ποια νομική βάση το δίνουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παρέμβουμε σε ατομικές περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να παρεύουμε στην ανεξαρτησία των δικαστικών συστημάτων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία για τους καταναλωτές, αλλά να έχετε υπόψη ότι η δικονομία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές, ιδιαίτερα δημιουργώντας, ε, ε, δημιουργώντας ευνοϊκούς ε, νόμους, κανόνες για τη δικαιοδοσία, κατά τα άλλα είναι ουδέτερη. Πρέπει να είναι ίδια για όλους δεν αφορά μόνο τις ε, καταναλωτές. Ο κύριος Βέλμπροκ είναι καταναλωτής. Άλλο άλλος είναι εμπορευόμενος. Η διαδικασία πρέπει να είναι ουδέτερη. Και ως ουδέτερη δεν είναι δυνατόν να ευνοεί τον καταναλωτή έναντι του ε, εμπορευομένου. Αυτή είναι η αστική δικονομία. Μπορεί να είναι χρήσιμη για τους καταναλωτές. Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του κέντρου καταναλωτών του Κιέλου, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει θαυμάσιους ε, συνεργάτες, αλλά τονίζω. Στην περίπτωση του κυρίου Βέλμπροκ δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι έγινε οτιδήποτε εσφαλμένα σε σχέση με τη διαδικασία, την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Αυτό που δεν έγινε σωστά είναι η εφαρμογή και σε κάθε κράτος μέλος. Ένα πράγμα είναι να υπάρξει μια απόφαση, το άλλο είναι η εφαρμογή της απόφασης. Συγγνώμη που επαναλαμβάνω κάτι. Σε κάθε διαμεθοριακή συναλλαγή ε, προκύπτουν ε, επιπλέον δυσχέρειες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει απόσταση. Μετά υπάρχει το γλωσσικό φράγμα. Αν το γερμανικό δικαστήριο ζητήσει κάτι από τον κύριο Βέρμπροκ, θα καταλάβαινε. Δεν θα είχε πρόβλημα. Ή κάποιο θα του έλεγε τι του ζητάει το δικαστήριο. Εάν λαμβάνει κάτι στα ισπανικά και χρησιμοποιεί αυτόματα συστήματα μετάφρασης, δεν καταλαβαίνει τη νομική ορολογία και επιχειρηματολογία. Αυτά είναι πρακτικά θέματα. Πολλοί θα θέλαμε να εφαρμόζονται όλες οι αποφάσεις. Όταν λαμβάνετε μία απόφαση πρέπει να εφαρμόζεται. Αλλά ακόμη και σε καθαρά ε, εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους δεν εφαρμόζονται πάντα όλες οι αποφάσεις. Αυτή η απόφαση για τον κύριο Βέλμπροκ αναγνωρίστηκε. Και έχουμε τα στοιχεία ότι το Ισπανικό Δικαστήριο είπε ναι θα εφαρμοστεί. Και μετά έχουμε στοιχεία ότι το Ισπανικό Δικαστήριο του είπε κατά ποιου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Και αυτό είναι πολύ ε, συνηθισμένη διαδικασία. Σε κανένα κράτος μάλλον δεν υπάρχει εξοφίκιο εφαρμογή. Πρέπει ο ενάγων να διασφαλίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί απόφαση, ότι θα εφαρμοστεί απόφαση. Και πρέπει να λάβετε υπόψη επίση ότι μπορείτε να λάβετε και νομική αρρωγή. Αν έχετε προβλήματα, θα πρέπει να επιχειρήσει να λάβει με βάση την οδηγία νομικής αρρωγής, νομική αρρωγή για διαμεθοριακές υποθέσεις. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειε της υπόθεσης. Σας περιγράφω το νομικό πλαίσιο. Ο κύριος Βέλμπροκ μπορεί να πάρει νομική βοήθεια από έναν Ισπανό δικηγόρο, ούτω ώστε να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Φυσικά, αν είναι δυνατόν να εκτελεστεί, γιατί μπορεί ο εμπορευόμενο κατά του οποίου εστράφει και κατά του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί, μπορεί να έχει πτωχεύσει και να μην υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιωθεί ο ενάγων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να πει σε κάποιον κάτι τέτοιο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι κάνουμε. Αναλύουμε τις λεπτομέρειες κάθε υπόθεση, αναλύουμε και τα οριζόντια θέματα. Γνωρίζετε τον πίνακα αποτελεσμάτων της δικαιοσύνης, που είναι μια προσπάθεια, ελπίζω επιτυχημένη, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, ρίξει μια ματιά στην ε, συγκεκριμένη λειτουργία των νομικών συστημάτων των κρατών μελών, των δικαστικών συστημάτων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να λάβουμε και να ε, επιτύχουμε να μας δίνουν στοιχεία με συγκεκριμένη μορφή. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία εξέτασε και συμπεριέλαβε ο πίνακας αποτελεσμάτων στοιχεία για την εφαρμογή των αποφάσεων. Ελπίζω έτσι η Κομισιόν να πιέσει και να οθήσει τα κράτη-μέλη να ε, βελτιώσουν τα δικαστικά τους συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξή τώρα. Όσον αφορά την αναφορά του κύριου Βέλμπροκ θα παραμείνει ανοιχτή. Θα συντάξουμε μια επιστολή προς τις Ισπανικές Αρχές ε, όπου θα τους ζητήσουμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα του συντομότερο δυνατόν. Και θα στείλουμε και μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν μπορεί να εκπονήσει κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά την άλλη αναφορά, αν κατάλαβα καλά, ο αναφέρον δεν έδωσε επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε την αναφορά. Οπότε τι θα κάνουμε, θα την κλείσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν την αναφορά 512 του κυρίου Βίτσε, διότι δεν περιλαμβάνει πληροφορίες επαρκής, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα. Οπότε κλείνουμε την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Έχω ίσχυ τη συνείδησή μου γιατί θα ανακοινώσουμε στον αναφέροντα γιατί κλείνουμε την αναφορά γιατί αν δεν μας ε, δώσει άλλες πληροφορίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αλλά μπορεί να μας στείλει άλλη αναφορά με άλλες πληροφορίες πρέπει να την κλείσουμε γιατί δεν έχουμε λάβει νέες πληροφορίες και θα το μάθει ο αναφέρον συμφωνώ λοιπόν Ωραία λοιπόν έτσι Αν έρθουν λοιπόν νέες πληροφορίες, πολύ φυσικά θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ένα νέο έντυπο και να ασχοληθούμε με την αναφορά αυτή ως νέα αναφορά. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα σε μια αναφορά ιταλική. Πρόκειται για την ε, αναφορά που αφορά το οικιακό εστιατόριο ως νέα ιταλική μορφή συνεργατικής οικονομίας. Πρόκειται για την αναφορά 1125 του 2016. Ο αναφέρον, ο κύριος Τζαμπατίστα Σιβολέτο, ελπίζω να το πρόφερα καλά, έχετε το λόγο κύριε Σιβολέτο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, ονομάζομαι Τζαμπατίστα Σιβολέτο. Και η αναφορά αυτή εστάλει από μια ομάδα επίδοξων ε, εστιατόρων Ιταλικών ε, ε, κατοίκων που σήμερα έχει 4.000 μέλη. Αφορά η home restaurant τους τομείς που βρίσκονται σε τεράστια ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας. Home restaurant σημαίνει ότι ανήκει στο σπίτι του και μαγειρεύει ε, οικογενειακά πιάτα, τοπικά πιάτα και διηγείται τις ιστορίες τους ε, στους ε, πελάτες. Απ' την άλλη, το να επιλέγει κανείς ένα home restaurant σημαίνει περιέργεια για να ανακαλύψει κανείς τις παραδόσεις ενός τόπου, την τοπική γαστρονομία που κληρονομείται από γονείς σε παιδιά, κάτι που είναι δύσκολο να βιώσει κανείς σε ένα κανονικό εστιατόριο. Μια τέτοια δραστηριότητα, όπως όλες οι δραστηριότητε που ενώνουν λαού και πολιτισμού, θα έπρεπε να έχει την ελευθερία να εκφραστεί και να αναπτυχθεί χωρίς πολλού δεσμού με την επιφύλαξη φυσικά του κανονισμού που να εμποδίζει ε, τυχόν στρεβλώσει. Στην Ιταλία όμω, μόλι οι πρώτε οικογένειε ξεκίνησαν να υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία των home restaurant, οι ενώσει τη κλασική εστίαση κατάφεραν να επιτύχουν από το Υπουργείο Οικονομική Ανάπτυξη μια γνωμοδότηση που εξισώνει τα home restaurant με τα κανονικά εστιατόρια. Με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν και που δεν συμβιβάζονται με μια δραστηριότητα που γίνεται σε ιδιωτικό χώρο. Ε, η, τα πρόστιμα των άνω των 10.000 ευρώ και η εκστρατεία ε, που μοιάζει με κυνήγη μαγισσών ουσιαστικά έχει καταπνίξει το φαινόμενο αυτό εν τη γενέση του και έχει αποθαρρύνει νέα ε, τέτοια εστιατόρια αναμένοντας να θεσπιστεί σχετική νομοθεσία. Το νομοσχέδιο για τα home restaurant που αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς μας ε, παραβιάζει τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Συνεργατική Οικονομία και αυτό εμπεβεβαιώνεται και από την ε, ε, αρχή εγγύησης του ανταγωνισμού και της αγοράς. Η επόμενη κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει την απαραίτητη διαδικασία, ωστόσο θα βρεθούν διάφορα εμπόδια όπως είναι και στην Ιταλία. Αυτή η ιδέα του Χόμπρεστονα που είναι πολύ όμορφη και απαραίτητη θα θέλαμε να ενθαρρυνθεί από εσά να την υπερασπίσετε ενώπιον του Ιταλού νομοθέτη, ώστε να αναθεωρηθεί η γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξη, που μπλόκαρε ουσιαστικά την ανάπτυξη αυτή τη πολλά υποσχόμενη δραστηριότητα ε, του sharing economy. Τέλος, ως Ευρωπαίος επιχειρηματίας θέλω να πω ότι αισθάνομαι ε, ότι μου απαγορεύεται να ε, πραγματοποιήσω τις δραστηριότητε που θα ήθελα, ενώ αυτό είναι δυνατό σε άλλες ε, χώρες. Και όλο αυτό έχει καθυστερήσει τις δικές μας προσπάθειε σε μεγάλο βαθμό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιβολέτο. Ο... Κύριε Γιάννη Στάιν, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσει. Πράγματι η κατοίκον μαγειρική, το home cooking είναι μια δραστηριότητα που ελκύει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές. Είναι μια από τις πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από μη επαγγελματικές πλατφόρμες. Αυτούς που ονομάζουμε ομότιμους, ανθρώπους που δεν λειτουργούν υπό επαγγελματική ιδιότητα. Όπως είπε ο Ναφέρον, έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση για τη συνεργατική οικονομία τον Ιούνιο του 2016, όπου επισημαίνουμε τη διαφορά μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από επαγγελματίες και υπηρεσιών που παρέχονται από μη επαγγελματίες, από ομοτήμους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιβολέτο που επεσήμανε το ζήτημα σε εμάς ε, ότι είμαστε ευγνώμονες. Μετά από την ενημέρωση που λάβαμε από τον αναφέροντα, ήρθαμε σε επαφή με τις Ιταλικές Αρχές ε, και συζητήσαμε το νομοσχέδιο. Οι επαφές αυτές ε, έκαναν τις Ιταλικές Αρχές να κοινοποιήσουν το νομοσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθησε μια περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μεταξύ, και πληροφοριών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των Ιταλικών Αρχών για το νομοσχέδιο. Ξέρουμε επίση ότι η Αρχή Ανταγωνισμού τη Ιταλία έχει εκδώσει μια γνωμοδότηση για το νομοσχέδιο νωρίτερα φέτο αναφέροντα ότι πιστεύει ότι αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λόγω τη επιβολή ε, αδικαιολόγητων περιορισμών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτέ τι επαφέ με τι Ιταλικέ Αρχέ. Εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όλε οι πλευρέ μπορούν να ακουστούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα συμμετέχει. Τώρα, σε περίπτωση που στο τελικά η Ιταλία αποφασίσει να υιοθετήσει ε, τέτοια νομοθεσία, τότε φυσικά, όπως ε, πάντα ως θεματοφύλακες των συνθήκων θα ε, αξιολογήσουμε την νομιμότητα της Ιταλικής νομοθεσίας ε, και κατά πόσο μορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα, θα βάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε αν υιοθετηθεί να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Ευχαριστούμε που θέσατε αυτό το θέμα υπόψη μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιβολέτο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα στα δικά μας μάτια είναι πολύ σημαντική. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ιταλία, αλλά οι νόμοι της Ιταλίας να αντίκεινται σε αυτή τη ε, διαδικασία. Ο κύριος Τσίριο έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την εστίαση, όπως και πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας μας πλέον. Διότι αυτό που βλέπουμε συγκρίνοντας τα home restaurant με τα κανονικά εστιατόρια, το βλέπουμε και συγκρίνοντας την Uber με τους ε, αυτοκινητιστές, με τους ανθρώπους που νοικιάζουν το σπίτι τους, ε, το εξοχικό τους σε τουρίστες, ε, σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία. Έχουμε μια κατάσταση δηλαδή που αφενός αποτελεί ε, σύμπτωμα μιας ε, οικονομίας που μεταβάλλεται παρέχοντας στους καταναλωτές πιο βολικές υπηρεσίες. Από την άλλη φυσικά μπορεί να ε, θέσει σε κίνδυνο συγκεκριμένα επαγγέλματα διότι το επάγγελμα του εστιατόρα είναι επάγγελμα όταν μιλάμε λοιπόν για εστίωση, μιλάμε και για υγειονομικούς κανόνες ε, πολύ συγκεκριμένους. Η γνωμοδότηση των Ιταλικών αρχών ουσιαστικά επιχειρεί να διασφαλίσει ότι όταν ένας καταναλωτής, ένας πολίτης πάει να φάει στο σπίτι κάποιου άλλου ιδιώτη, στο σπίτι αυτό θα τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες ε, μεταξύ άλλων που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του εν λόγω καταναλωτή. Χωρίς να ξεχνάμε και τις φορολογικέ πτυχές, διότι είναι προφανέ ότι σήμερα ενώ η Ιταλική φορολογία για ένα εστιατόριο, για οποιαδήποτε επιχείρηση κυμαίνεται στο 50 με 60%, ε, παραλαμβάνω 57 με 60%. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει κάποιος δηλαδή 8 μήνες ε, το χρόνο για το κράτος και τέσσερι μήνε για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και ξαφνικά να υπάρχουν στην αγορά προσφορέ που θα φορολογούνται πολύ χαμηλότερα αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό. Παρότι λοιπόν ναι, πράγματι το home restaurant είναι μια συναρπαστική δραστηριότητα επικοινωνίας ε, και καταπληκτική υπηρεσία ε, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα διότι τέτοια επαγγέλματα ε, χρήζουν προστασίας. Η Ιταλία έχει γίνει γνωστή χάρη στους σεφ, στους μάγειρους της, ε, στους μαγειρούς της, στα, ο φαγητό της. Ναι, βασίζεται όλο αυτό στην οικιακή παράδοση, στο πώς μαγειρεύαν οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, αλλά οι εστιατόρες είναι αυτοί που έκαναν γνωστή τη χώρα μας. Οπότε, ναι, πολύ ωραίο το επιχείρημα να είμαστε ανοιχτοί στα καινούργια πράγματα. Απ' την άλλη, όμως, να μην ξεχνάμε ότι όσοι ασκούν αυτό το επάγγελμα εδώ και γενιές πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτερ. Ναι, να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Είναι πολύ σωστά. Και το βασικό είναι να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει ένα όριο υπάρχει κίνδυνος εάν ε, γίνουν επιχειρήσεις στα σπιτικά εστιατόρια να κινδυνεύσουν τα άλλα εστιατόρια. Δεν υπάρχει βέβαια νομοθετική βάση, αλλά οι κυρώσεις είναι βέβαια ταχείες. Θα μπορούσε κάθε κράτος να ε, υιοθετήσει κάποιους νόμους. Βεβαίως θέλουμε να μπορούμε να πάμε να φάμε κάπου, αλλά ε, δεν πρέπει να θέσουμε εν κινδύνο τον κλάδο της εστίασης. Δεν ξέρω. Μπορούμε να πούμε στους Ιταλούς να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, να πείτε τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Δεν θέλουμε να πνίξουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες χωρίς να θέσουμε εν κινδύνο τον κλάδο. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι υπάρχει το πρόβλημα με την ε, ενοικίαση ιδιωτικών ε, κατοικιών ε, σε φίλους ή γνωστούς. Τι είναι φίλος και γνωστός, ε, πού χρειαζόμαστε και πού δεν χρειαζόμαστε νομοθετικές ρυθμίσεις. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι πάντα πιο καινοτόμα από τους νόμους, αλλά ο νόμος εκ των υστέρων πρέπει να διορθώνει την κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι ο αναφέρον εκνευρίζεται που δεν υπάρχουν σαφείς νόμοι, αλλά βεβαίω οι κυρώσεις έρχονται γρήγορα ενώ νόμοι καθυστερούν. Οπότε απευθύνομαι στους συναδέλφους. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να παρακαλέσουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει σύντομα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, στρέφομαι προς τους συναδέλφους. Εσείς ε, που ξέρετε την κατάσταση, τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την αναφορά. Πίτερ, παρατηρούμε ότι στην Ιταλία κάτι τρέχει σε νομοθετικό επίπεδο επίσης. Παρατηρούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Ιταλικές Αρχές. Υποστηρίζουμε τέτοιου είδους επικοινωνία και θα πρέπει να αναμένουμε να ολοκληρωθεί. Οπότε αφήνουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και θα την ξαναδούμε σε μερικούς μήνες κύριε Σιβολέτο όταν θα έχουμε νέες πληροφορίες από την Ιταλία. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Το τελευταίο μας ε, θέμα επίσης είναι μια Ιταλική αναφορά. Ε, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για την ε, διακριτική φορολογία για τον τομέα της τρούφας στην Ιταλία και της τρευλώσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο κύριος Μάριο Καρμπόνε είναι ο αναφέρον, βρίσκεται εδώ μαζί μας, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους Επιτρόπους και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Έχουμε ξανασυζητήσει και το επιχείρημα αυτό και ήταν αποτελεσματική συζήτηση. Ήταν το να ασχοληθούμε με το θέμα του τρούφας από φορολογική και ρυθμιστική άποψη ουσιαστικά να εξισωθεί ε, στην Ιταλία η, νομοθεσία της Ιταλίας με εκείνη των άλλων χωρών. Η Ιταλία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ε, λευκής τρούφας σε σχέση με τη μαύρη, σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχει πολύ λευκή τρούφα ε, μη καλλιεργημένη ουσιαστικά φύεται φυσιολογικά και αυτό έχει δημιουργήσει σε διάφορα προβλήματα τόσα χρόνια γιατί δεν έχει ουδέποτε αντιμετωπιστεί ως γεωργικό προϊόν. Οι τρούφες ε, φύονται σε μέρη όπου υπάρχουν κυρικές δραστηριότητες που ευνοούν το περιβάλλον, παρότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καλλιέργεια αυτή καθεαυτή. Έτσι λοιπόν σε φορολογικό επίπεδο αντιμετωπιζόταν ανέκαθεν όχι σαν γεωργικό προϊόν, με συνέπεια να φορολογείται και σε επίπεδο ΦΠΑ ε, δυσμενός σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίε αυτή τη Επιτροπή ήταν πολύ αποτελεσματικέ, διότι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η Ιταλία αναγκάστηκε να προσαρμόσει το σύστημα ε, ΦΠΑ ε, σύμφωνα με αυτό που ισχύει στι άλλε χώρε. Οπότε ευχαριστώ για την παρέμβασή σα και τι άλλε χώρε, Αλλά παραμένει το δεύτερο πρόβλημα, ότι δεν πλαισιώνεται ω γεωργικό προϊόν. Το γεγονό ότι δεν είναι γεωργικό προϊόν δημιουργεί δύο μεγάλε δυσκολίε. Η πρώτη είναι φορολογική. Τα γεωργικά προϊόντα φορολογούνται λιγότερο, έχουν πιο ευνοϊκή φορολογία όπω είναι φυσιολογικό σε όλε τι χώρε ε, τη Ευρώπη. Οπότε Πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η φορολογία ώστε το προϊόν αυτό να γίνει ανταγωνιστικό για τις επιχειρήσεις μας όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο ζήτημα είναι πιο σοβαρό όμως. Οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή δεν είναι γεωργικό προϊόν είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί σε όλες ε, ε, της δράσης ε, στήριξης της γεωργίας ε, προβλέπονται στην Ευρώπη. Οπότε δεν εντάσσονται σε όλα αυτά τα προγράμματα στήριξης οι τρούφες, διότι δεν είναι γεωργικά προϊόντα, οπότε δεν ξέρουμε αν πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τη γεωργία ή από τα κονδύλια που καλύπτουν τη δασοκομεία. Βρίσκονται δηλαδή σε ένα νομικό ε, χάσμα μεταξύ δύο τομέων. Οπότε μειώνεται η παραγωγή, εγκαταλείπονται σιγά σιγά τα εδάφη ε, αυτά της δασοκομείας, οπότε έχουμε μια υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, προβλήματα υδρολογικά, διότι κάθε δάσος που εγκαταλείπεται αποτελεί κίνδυνο όταν ε, πέφτουν τα νερά και μετά είναι που μειώνεται και υποβαθμίζεται η παραγωγή. Η λευκή τρούφα είναι ένα από τα πιο αγαπητά προϊόντα στην Ευρώπη και στην Ιταλία. Ε, χρησιμοποιείται στην εστίαση υψηλού επίπεδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει οπωσδήποτε να τη διασώσουμε ω προϊόν και γι' αυτό απαιτούνται καθαρά γεωργικέ πολιτικέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και αν στη δυνατόν η Ιταλική ε, κυβέρνηση να εντάξει τη λευκή τρούφα στα γεωρικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα στου επόμενε μήνε, γιατί αυτή τη στιγμή συζητείται μια τροπολογία ε, στην νομοθεσία προπολογισμού που μπορεί να αφορά είτε το δημοσιονομικό είτε το γεωργικό κομμάτι και δεδομένη τη αποτελεσματικότητα τη δική τη Επιτροπή στα θέματα ΦΠΑ, ε, ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ώστε να κλείσει επιτυχώ η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Καρμπόνε. Για την Κομισιόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ταξινόμηση των διαφόρων ειδών τρούφας στην ε, συνδυασμένη ε, ονοματολογία. Έγινε αντικείμενο ανάλυση και καταλήξαμε ότι και από την πλευρά του παραρτήματος 1 της ηθίκης που καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και με βάση την ε, δική μας κοινή οργάνωση αγοράς 1308 του 2000 16. Με, 13. Με βάση το εναρμοσμένο σύστημα όσον αφορά οι τρούφες υποπίπτουν σε δύο διαφορετικά κεφάλαια. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά κεφάλια και με βάση το δικό μας κανονισμό και με τη συνθήκη 1308-2013 καλύπτονται οι τρούφες. Και στο σημείωμά μας αναφερόμεθα αναλυτικά στους αριθμούς στην ονοματολογία για τις διάφορες ε, τρούφες. Καλύπτονται όλες τα διάφορα κεφάλαια. Παράδειγμα έχουμε ένα κεφάλαιο για τα εδόδημα, λαχανικά και ρίζες. Και ένα άλλο κεφάλαιο καλύπτει τα μεταποιημένα λαχανικά, τα εδέσματα από λαχανικά. Και σε αυτές τις δύο κατηγορίες αναφέρονται οι τρούφες. Από πλευράς λοιπόν συμπερίληψης Οι τρούφες είτε είναι νοπές είτε έχουν υποστεί κατεργασία καλύπτονται από την νομοθεσία μας. Αυτά είναι τα... Αυτά είναι... Αυτά είναι αυτά που προκύπτουν από την ονοματολογία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο. Εσείς παρακαλώ. Ο κύριος Σύριο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ήθελα να επισημάνω ότι οι εργασίες που κάνουμε εμείς εδώ τελικά χρησιμεύουν. Όπως υπενθύμισε προηγουμένως και ο αναφέρον μάλιστα, Εμεί ε, επ' αυτής της αναφοράς έχουμε επιτύχει ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα διότι το ΦΠΑ για την τρούφα στην Ιταλία έπεσε από το 22% σήμερα στο 10%. Και αυτό συνέβη ε, και χάρη στη δική μας καταγγελία που έγινε εντός της Κομισιόν ε, και οι επαφές που ακολούθησαν με την Ιταλική κυβέρνηση η οποία προσάρμοσε στη συνέχεια την, το ΦΠΑ για την ε, τρούφα σύμφωνα με τις άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Η μισή δουλειά έγινε λοιπόν. Ε, η άλλη μισή δουλειά είναι να βάλουμε την τρούφα στην κατηγορία που ανήκει. Εάν σε όλη την Ευρώπη, αν κατάλαβα καλά εγώ τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, εάν ολόκληρη η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας λέει ότι η τρούφα είναι γεωργικό προϊόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ιταλία, όντας μέσα στην Ευρώπη, μπορεί να συνεχίσει να ορίζει την τρούφα ως νομικό κενό. Δηλαδή ως αρεσνούλιους, ως ε, ένα αντικείμενο ε, το οποίο φύεται ε, μόνο του και αποτελεί διοκτησία όποιου το βρει. Τώρα, δεδομένου ότι η τρούφα είναι ένα μανιτάρι που μεγαλώνει κάτω από τη γη, Άλλε κατηγορίες όπως τα μανιτάρια, τα πορτσίνη θεωρούνται ε, γεωργικά προϊόντα που φύονται από μόνα τους. Η διαφορά τους με τα καλλιεργημένα είναι ότι αυτά που φύονται μόνα τους μπορεί κάποιο να πάει να τα βρει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ιδιοκτήτη ε, οικοπαίδου. Ο ιδιοκτήτη, μάλλον του οικοπαίδου, δεν είναι ιδιοκτήτη του προϊόντο αυτού. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πάω να πάρω με να, να μαζέψω κεράσια από το δένδρο ε, κάποιου αγρότη, αλλά μπορώ να πάω να μαζέψω τα μανιτάρια, γιατί είναι αυτοφύη που βρίσκονται κάτω από το κερασιά. Αφού είναι αυτοί οι κανονισμοί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, και αφού τα καταφέραμε και με το ΦΠΑ, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γράψει τι Ιταλικέ Αρχέ, επισημένοντα το πρόβλημα και εκφράζοντα την επιθυμία να ε, διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να υπάρχει ομοιομορφή αντιμετώπιση του προϊόντος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκινάσκη θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ασχολήθηκα εγώ προσωπικά με τις καταγγελίες που έλαβε η Κομισιόν. Ε, ξεκινήσαμε διαδικασίες EU Pilot ε, και διάλογο με την Ιταλία και πράγματι επιτύχαμε μια σημαντική νομοθετική αλλαγή με μείωση του ΦΠΑ. Τώρα, σε σχέση με το κατά πόσον οι τρούφες είναι ή δεν είναι γεωργικό προϊόν, η θέση της Κομισιόν, το ακούσατε, είναι πως πρόκειται για γεωργικό προϊόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, ενδεχομένως υφίσταται μια παρερμηνία. Ο στόχος ήταν να αναγνωρίσουν οι Ιταλικές αρχές ότι ε, οι τρούφες είναι γεωργικό προϊόν προκειμένου να αλλάξει το φορολογικό καθεστώ και να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι πλέον στο 10% και έχω την εντύπωση ότι ο στόχο θα ήταν να μειωθεί στο 4% που είναι ο ε, ΦΠΑ για τα γεωργικά προϊόντα ή 5% ε, που είναι ένας καινούριος φορολογικός συντελεστής που εισήγαγε τελευταία Ιταλία. Ε, σύμφωνα με την οδηγία ΦΠΑ, τα κράτη-μέλη γνωρίζετε ε, έχουν δικαίωμα να διαθέτουν δύο μειωμένους φορολογικούς συντέλεστες ΦΠΑ συν την δυνατότητα διατήρησης έναν, ενός υπερχαμηλού, υπερμειωμένου συντελεστή υπό την προϋπόθεση ότι αυτός υφίστατο ήδη την 1η Ιανουαρίου 2011. Ε, 1991. Τότε στην Ιταλία υφίστατο συντελεστής 4%. Τώρα, που βρίσκεται. Το γεγονός ότι ένα προϊόν θεωρείται ε, γεωργικό ή όχι δεν επηρεάζει στην πράξη τον συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος θα εφαρμόζεται σε αυτό. Διαβάζοντας την Ιταλική νομοθεσία θα δούμε ότι υπάρχουν γεωρικά προϊόντα τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 10% ΦΠΑ. Συνεπώς, αν αύριο η Ιταλία να γνωρίσει την τρόφο ως γεωργικό προϊόν δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή 4%. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αυτοματισμός. Η Κομισιόν θα έπρεπε να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση αν ε, η Ιταλία εφάρμοζε το συντελεστή 4%. Η οδηγία το απαγορεύει. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ιταλία είναι να εφαρμόσει συντελεστή 5% που είναι ένα συντελεστή ο οποίος πρόσφατα εισήχθη ε, για την φορολόγηση του ριζότο, του βασιλικού και της ε, σάλβιας, της φουβασκόμηλου. Η Κομισιόν δεν ε, έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει όμως την Ιταλία να μειώσει ακόμα περισσότερο το συντελεστή ΦΠΑ της τρούφας στο μέτρο που τα κράτη-μέλη έχουν μια σημαντική φορολογική ανεξαρτησία ως προς αυτό το ζήτημα. Η αρχή της ουδετερότητας χαρακτηρίζει την οδηγία ΦΠΑ. Σύμφωνα με αυτήν, ε, παρόμοια προϊόντα, ισοδύναμα προϊόντα, πρέπει να την χάνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης στην πράξη δηλαδή, να υπόκειται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τρούφα, δεν είναι προφανές, δεν είναι ξεκάθαρο ότι ε, ο μέσος καταναλωτής θεωρεί την τρούφα ισοδύναμο συγκεκριμένων τύπων ε, μανιταριών. Ε, πιο μάλλον θα θεωρεί ο μέσος κατανοητής την τρούφα ένα προϊόν πολυτελείας, delicatessen και η Κομισιόν δεν είναι εύκολο να καταρρύψει την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποδίδει ένα μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας. Ελπίζω να σας διευκρίνησα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που είπατε ό,τι ήταν δυνατό, ό,τι και δεν είναι δυνατό σε σχέση με αυτό το θέμα που βρίσκονται τα όρια. Σημειώνουμε όλα αυτά που ακούσαμε. Είναι σημαντικό για τον ε, αναφέροντα ο κύριος Σύριο Μα πρότεινε να απευθύνουμε μια επιστολή στι Ιταλικέ αρχέ Ούτω και θα πράξουμε και θα δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ιταλία στο άμεσο μέλλον. Διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά και θα επανέλθουμε σε μερικού μήνε. Συμφωνείτε, κύριε Τσίριο. Ναι, να σας ευχαριστήσω. Να επισημάνω μόνο ένα πράγμα. Την Ιταλία δεν την ενδιαφέρει να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ. Δεν είναι τίθε θέμα ΦΠΑ. Το θέμα είναι ότι εάν ένα μήλο είναι φρούτο και αν ένα σολομός είναι ψάρι, ε, η τρούφα είναι γεωργικό προϊόν. Και μετά το ΦΠΑ είναι το αποτέλεσμα. Αλλά αν στις Βρυξέλλες η τρούφα θεωρείται γεωργικό προϊόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θεωρείται γεωργικό προϊόν και στην Ιταλία. Αυτό είναι το παράλογο. Δεν είναι φορολογικό το θέμα. Η Ιταλία θα αποφασίσει ποιο ΦΠΑ θα επιβάλλει ούτω ή άλλω. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Το θέμα μα είναι ότι αν το μήλο θεωρείται μήλο Βρυξέλλες και θεωρείται και φρούτο και γεωρικό προϊόν, αν θεωρείται γεωρικό προϊόν στις Βρυξέλλες πρέπει να θεωρείται γεωρικό προϊόν και στη Ρώμη. Αυτό είναι το θέμα. Πού κατατάσσεται δηλαδή το προϊόν. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ωραία, θα γράψουμε λοιπόν αυτή την επιστολή στις Ιταλικές Αρχές. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε ένα διάλογο με τις αρχές αυτές και θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Και θα επανέλθουμε αργότερα στο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα εργασιών μας. Επιτρέψτε μου, πριν κλείσω τη συνεδρίαση, να σας πω κάτι το σημαντικό. Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία μας συνεδρίαση ε, φέτος της Επιτροπής μας. Ε, σύμφωνα με την δική μου αξιολόγηση και με τη γενική αξιολόγηση, η Επιτροπή Αναφορών έκανε σημαντική εργασία κατά τη διάρκεια του 2017. Ασχοληθήκαμε με θέματα πραγματικά ουσιώδη, ευαίσθητα, επίγοντα και Είχαμε μια θαυμάσια ομάδα με την οποία εργαστήκαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Πέτερ, εσύ εκπροσωπεί όλους του συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μας, ε, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων. Από πλευράς της ε, κυρίας Προέδρου, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ε, καλές γιορτές θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας τον Ιανουάριο.